Colleagues, con I, I would like you to... Συνάδελφοι, παρακαλώ. Επιτρέψτε μας να συνεχίσουμε με επεξηγήσεις ψήφου. Παρακαλώ, αποχωρήστε ησύχως. και με φταξιά. Începem, trecem la explicațiile Λοιπόν, περνούμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι μπορείτε επίσης να καταθέσετε επεξηγήσεις γραπτός. Έχουμε 50 συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να λάβουν τον λόγο. Σας παρακαλώ λοιπόν να τηρήσετε αυστηρό τον χρόνο του ενός λεπτού. Ο κ. Πόσπισιλ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, για το σύστημα ηλεκτρονικής ειδοποίησης περιπτώσει εκτάκτου ανάγκης επιοχημάτων δεν μπόρεσα να ψηφίσω διότι η κάρτα μου δεν λειτουργούσε. Θα το πράξω αργότερα. Θα ψηφίσω όμως κατά εκ μέρους της Άλντε. Παρά το γεγονό ότι είμαι υπέρ αυτού του συστήματο του οικόλυπη οχημάτων. Ε, δυστυχώς δεν ψήφισα λόγω του ότι δεν λειτουργούσε η κάρτα μου. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Κυρία Μπιλιάνα Μπορσάν, ένα λεπτό. Μιλιάνα Μπόρζαν, παρακαλώ. Δεν είναι στην αίθουσα. Μάρκους Πίπα. Δόμνα Μλίνα Ραγγέλικα. Η Νταμναρίνα Αναγγέλικα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, κοιτάξτε, εγώ ε, μία πρόταση και υπερψήφισα ε, βεβαίως και εγώ είμαι υπέρ της μεγαλύτερης ε, ασφάλειας στις οδικές μεταφορές, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να μην θυσιάζουμε κάθε φορά την ελευθερία μας. Είτε πρόκειται για την ε, συλλογή δεδομένων, είτε πρόκειται για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, όταν πρόκειται για το e-call, πάντα εμείς είμαστε υποποίηση και εγώ ως ελεύθερος άνθρωπος διαφωνώ το σύστημα αυτό το e-call υποτίθεται θα δώσει τη δυνατότητα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν υπάρχει ατύχημα να προσφέρεται ταχύτατα βοήθεια αλλά όπως ε, και πολλοί άλλοι και εγώ φοβάμαι ότι αυτό το σύστημα απλά θα βοηθήσει στο να μας παρακολουθούν συνέχεια και με τον τρόπο αυτό να διεισδύουν στην ιδιωτική μας σφαίρα. Όταν ακούω ότι πρόκειται για ένα σύστημα ενυπνώση όπου έτσι κι αλλιώς όλα θα σβήνονται, ε, σε μένα χτυπάει αυτό ένα καμπανάκι γιατί και ένας ε, τίγρης εν υπνώση είναι ένας κοιμόμενος τίγρης. Γιατί λοιπόν δεν μπορεί κανείς να δώσει τη δυνατότητα επιλογής στους πολίτες, δηλαδή το να ανοίγει ή να κλείνει κανείς το σύστημα, κατά το δοκούν, εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ο κύριος Πίκουλα για ένα λεπτό. Πάρα πολλοί άνθρωποι ε, χάνουν τη ζωή τους ε, στους δρόμους, ε, οι αριθμοί σοκάρουν και γι' αυτό το λόγο πρέπει να απαντήσουμε. Το e-call είναι μια χρήσιμη υπηρεσία, μπορεί να βοηθήσει κάθε λεπτό που σώζουμε έναν άνθρωπο αυτό ή μάλλον κάθε λεπτό που εξοικονομούμε βοηθούμε έναν άνθρωπο να σωθεί. Και ελπίζω βεβαίως σε αυτό το σύστημα να εντάσσονται και οι αρχές της προστασίας των δεδομένων. Οι τεχνικές προτάσεις είναι καλές και έχουμε αρκετό χρόνο για να εισάγουμε το σύστημα Γι' αυτό και εγώ ε, το στηρίζω ανεπιφύλακτα και συγχαίρω τον εισηγητή που εργάζεται πάνω στο θέμα εδώ και δύο θητείες. Νομίζω λοιπόν ότι έχει φτάσει πια η χρονική στιγμή να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα μπορεί να σώσει μέχρι και 2.000 ζωές το χρόνο. Πρέπει να εισαχθεί το σύστημα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ο κύριος Νέκοβ. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή ή την εισηγήτρια για τα ε, για την έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να διασφαλίσει το σύστημα αυτό, να είναι σίγουρη πριν εισαχθεί σε πολλά αυτοκίνητα το 2018. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ως προς την ασφάλεια των πολιτών της και γι' αυτό πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει ταχύτατα να εφαρμόσει τα μέτρα που θα επιτρέψουν ε, την ε, τοποθέτηση αυτού του συστήματος. Η υπηρεσία θα πρέπει να είναι ε, προσπελάσιμη και εύχριστη για όλους τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Πάνω από 20 τόσες χιλιάδες άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο στους δρόμους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τι να κάνουμε, να περιμένουμε και άλλα χρόνια να είναι υποχρεωτική αυτή η ζωή τη στιγμή που μια ζωή είναι χαμένη. Ο κύριος Μαριάς παρακαλώ, για ένα λεπτό την τεράστια χρησιμότητα ενός συστήματος όπως το ecall το οποίο θα μπορέσει πράγματι να σώσει ζωές μετά από τροχαία ατυχήματα. όμως το ecall δεν παρέχει εγγυήσεις για τη διασφάλιση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής και αυτό διότι πρώτον το ecall εγκαθίσταται υποχρεωτικά σε όλα τα αυτοκίνητα δεύτερον θα συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και παρά τη θέληση του οδηγού τρίτον γιατί με την αρχή της ευελιξίας δημιουργούνται σημαντικά κενά στην προστασία της ιδιωτικής ζωής τέταρτον διότι τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για κάποιο χρονικό διάστημα πέμπτον διότι τα προσωπικά δεδομένα θα είναι στη διάθεση ιδιωτικών φορέων. επομένως το σύστημα ecall θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση του μεγάλου αδερφού που επιχειρεί να ελέγξει κάθε πτυχή της ιδιωτικής μας ζωής. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή και θέλω να πω ότι δεν μπόρεσα να ψηφίσω την τροπολογία γιατί η κάρτα μου δεν λειτουργούσε. Δεν το ξέρα πριν ε, ζητήσω επεξήγηση ψήφου. Θέλω να πω λοιπόν ότι στηρίζω βέβαια το σύστημα, έχω όμως παρόλα αυτά και κάποιες ανησυχίες. Πολλά επόθηκαν για τα δεδομένα τα οποία διατηρούνται. Επειδή υπάρχει αρχή του συστήματος Dorman, θέλω να τονίσω το οποιοδήποτε σύστημα το οποίο διατηρεί δεδομένα για μια συγκεκριμένη περίοδο μπορεί να τύχει κατάχρησης. Η τεχνολογία, πρόοδος προχωρούν πολύ γρήγορα. Μερικές φορέ δεν μπορούμε να προβλέψουμε κατά πόσο θα γίνει ή δεν θα γίνει κατάχρηση του συστήματος. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα ένα σύστημα το οποίο να μπορεί κανείς να κλείσει, να εξουδετερώσει αν θέλει. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό τώρα κύριε Χάρκεν. Στηρίζω την τροπολογική για το e-call. Προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στα προσωπικά, την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και το κοινό καλό. Πρέπει να δούμε στην περίπτωση τέτοιων συστημάτων πώς θα προστατεύσουμε τα δεδομένα, αλλά από την άλλη μεριά μην ξεχνάμε ότι σώζουμε ζωές και χρήματα. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν στηρίζω την τροπολογία που προτάθηκε και που λέει ότι οι κατασκευαστές πρέπει να διασφαλίσουν ότι μπορεί ο χρήστης να κλείσει το σύστημα με το χέρι. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει να έχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στον ιδιωτικό βίο και συγχρόνως να σώζουμε ζωές. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ρήτρες ασφαλείας, ότι δεν θα μπορεί κανείς πριν συμβεί ατύχημα να εντοπίσει τον χρήστη και ότι τα, δεν θα παρακολουθούνται τα δεδομένα. Τα κέντρα κατεπήγοντος δεν θα μπορούν χωρίς να υπάρχει ρητή συνένεση του χρήστη να μεταφέρουν δεδομένα. Χαίρομαι που υπάρχει αυτή η προστασία. Ευχαριστούμε κύριο Γιάρ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι σήμερα είναι μια πολύ καλή ημέρα για την ασφάλεια των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το σύστημα αυτό ολοκληρώνουμε τη στρατηγική μας. Ε, παλαιότερα είχαμε έναν ενιαίο ρυθμό για πρώτες βοήθειες. Τώρα έχουμε το σύστημα Είναι πολύ σημαντικό να εγκατασταθεί σε όλα τα αυτοκίνητα και ε, σε περίπτωση ανάγκης να τίθεται σε λειτουργία αυτόματα. Κρίμα που υπήρξαν μερικοί που διαφωνούν. Να αναγνωρίσουν το λάθος τους ε, και να σκεφτούν ότι όταν υπάρχει ατύχημα ε, και είναι πολύ μες στο αυτοκίνητο, ποιο θα αναλάβει να ενεργοποιήσει το σύστημα. Δεν νομίζω ότι θα θέλει κανείς να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θέλω να πω ότι πολύ σωστά υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο ε, επόμενο ομιλητή, ο κύριο Κέλλη, για ένα λεπτό. Εγώ θέλω να σας εξηγήσω ότι υπερψήφισα και χαίρομαι που ε, υπερψηφίστηκε η έκθεση. Βεβαίως ε, μετά από όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στους δρόμους Ευρωπαϊκής Ένωσης που πεθαίνουν 20 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει μιλάμε για κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια το χρόνο ε, αυτά τα στοιχεία πλήττουν και τη δική μου τη χώρα και ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ανθρώπους ε, οι οποίοι πεθαίνουν στους δρόμους, ε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η τεχνολογία e θα βοηθήσει. Όλοι πιστεύουμε ότι η πρόσβαση στον ε, χώρο του ατυχήματος θα είναι πολύ πιο γρήγορη, τουλάχιστον κατά 40% από ό,τι συμβαίνει τώρα. Και αυτό σίγουρα θα βοηθήσει στο να λυθεί το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ο κύριος ε, Κόσ για ένα λεπτό. Κυρία Σενάλοβα, εμείς ε, είμαστε, πήγαμε, προχωρήσαμε σε μεγάλο βαθμό μαζί. Το e είναι το μωράκι μας και σας ευχαριστώ πολύ που δεν παρασυρθήκατε από αυτούς που έχουν ε, επιφυλάξει. Αυτό το e βασίζεται στον αριθμό πρώτων βοηθειών που υπάρχει, το 112 νομίζω και μετά από κάποια χρόνια θα είναι υπεπατημένοι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ακόμα και τα φορτηγά και οι μοτοσυκλέτες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα και να σώζονται και μέχρι να γίνει αυτό λείπει ένα μικρό βηματάκι το να υπάρχουν τροχαία ατυχήματα με βαριά τραυματισμένος είναι εκείνο που μας οδήγησε στο να υποστηρίζουμε το σύστημα e-call. Επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ε, θέλω να πω ότι εγώ είμαι υπέρ της ε, οδηγίας ε, ECOL γιατί πιστεύω και αυτό αποδείχτηκε και από τη συζήτηση ότι για το μέλλον χρειαζόμαστε καλύτερη υποστήριξη και επίσης ε, πρέπει να περιορίσουμε την υποστήριξή μας ε, προς ε, εκείνα τα καύσιμα που βλάπτουν το περιβάλλον. Είμαι λοιπόν ευχαριστημένος που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε την πολιτική της ε, και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι μια παρεμφερή συζήτηση διεξάγεται τώρα στο Κοινοβούλιο της ε, Τσεχίας με αντικείμενο το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Και λυπάμαι πάρα πολύ που η συζήτηση στην Τσεχία είναι διαφορετική από τη, δική μας. Ελπίζω οι Τσέχοι να μιμηθούν αυτό που ε, θα κάνουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησε πάλι να εγκρίνει οδηγίε τεχνοκρατών εξαιτία τη ιδεολογία για τους τραγονάνθρωκες που οδηγούν σε αποψήλωση στην Ασία. Οι οικολόγοι μας θέλανε να καταργήσουν όλους τους τραγονάνθρακες στην Ευρώπη. Αυτό όμως που δεν έχουν καταλάβει ούτε, ούτε οι οικολόγοι ούτε οι μη κεμιδικέ οργανώσεις είναι ότι μάλλον ζημιά κάνουν. Ευτυχώς οι χώρε μέλη έχουν καταλάβει ότι μπορούν από μόνε του να υποστηρίξουν τα συμφέροντα των πολιτών τους και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει τις φιλοδοξίες της και τα χρήματα τα οποία επενδύονται στην πρώτη γενιά ανθρώπων να μην χαθούν και να σωθούν πολλές χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Έτσι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε ένα know-how το οποίο θα διευκολύνει την μεταφορά σε πιο προηγμένα βιοκαύσιμα. Ευχαριστούμε. Πόλτσακ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την ψηφοφορία αυτή για να τροποποιηθεί αρκετή Οδηγία 2009 28. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για μένα η ψηφοφορία αυτή ήταν δύσκολη. Πρώτον, δεν υποστηρίζω τα δύο βιοκαύσιμα που θα αναφέρονται ως συμβατικά, πρώτη γενιά δηλαδή, που επηρεάζει τη χρήση γης. Και εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι ε, ξέρουμε ποιε θα είναι οι συνέπειε συνολικά. Τελικά όμω αποφάσισα να τη στηρίξω την πρόταση αυτή. Διότι μειώνεται ο αρχικό στόχο και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, γιατί έτσι λαμβάνουμε υπόψη μα πώ χρησιμοποιούμε τη γη μα και τι αφήνουμε στι επόμενε γενιέ. Πάντω, εγώ δεν θα ήθελα μελλοντικέ προσπάθειε με υπερφιλόδοξου στόχου που να συνοδεύονται από μη κριτική άποψη του πώς θα επηρεάσουν ε, την χρήση γης και τις επόμενες γενιές ε, κάθε απόφασή μας. Η ε, κυρία Χαρκίν στήριξα την οδηγία αυτή, αλλά καθαλό παρά ιδανική είναι. Πιστεύω ότι αντιμετωπίζουμε τα αρνητικά των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιοκαύσιμα και κυρίως τις επιδοτήσεις που γίνονται. Προωθούμε την ανάπτυξη προηγμένων βιοκαυσίμων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πέτυχε πολλούς από τους στόχους του, όμως ο συμβασμός αυτός θα διασφαλίσει θετικά για τις επόμενες γενιές. Οι χώρες μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να βάλουν τους δικούς τους ε, στόχους και όρια και επίσης θα πρέπει να δίδονται στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τους παραγωγούς και θα ληφθούν υπόψη και εκπομπές ILUC για τα βιοκαύσιμα στο μέλλον. Επιπλέον, οι ενεργειακές εισοδιές θα συμπεριληφθούν στην περικοπή του 7%. Δεν είναι τόσο φιλόδοξη η απόφαση αυτή όσο θα θέλαμε, αλλά είναι θετική. Ο κύριος Γιάρ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Τα βιοκαύσιμα τα επικρίνουμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των εισαγωγών που η παραγωγή τους δεν γίνεται βάση βιώσιμων μεθόδων. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε αυτήν την παραγωγή αμέσως, μιλάμε για μείωση 7%. Έχουμε θέσει στόχους όσον αφορά τις εκπομπές και ένα μέρος της παραγωγής πρέπει να έρχεται από τη δεύτερη-τρίτη γενιά βιοκαυσίμων. Πιστεύω πως με την εφαρμογή του κανονισμού αυτού πρέπει να αναρωτηθούμε πώς τα μέτρα αυτά τελικά θα έχουν θετικές επιπτώσεις στις τρίτες χώρες. Έχω τις αμφιβολίες μου. Πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει και μετά το 2020, γιατί χρειαζόμαστε ασφάλεια επενδύσεων για τη βιομηχανία. Ευχαριστώ. Πέτρι, λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ήδη είπα ότι θέλω η Ευρώπη να προωθεί πολιτικές τον οποίο στόχος είναι λιγότερη ρήπανση, καλύτερο περιβάλλον. Είμαι περήφανη που συμμετέχω σε μια κοινωνία η οποία είναι πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο και που υλοποιεί τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις της εν ώψη της συνάντησης των Παρισίων το κείμενό μας βαίνει προς την σωστή κατεύθυνση. Η ευθύνη μας ως συνομοθέτου είναι να αναγνωρίσουμε τους συμμάχους, μας, συμμάχους μας στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου. Πρέπει όμως να θέσουμε σαφείς στόχους και προθεσμίες να πούμε στη βιομηχανία, στους εργαζομένους, τι περιμένουμε από αυτούς να πράξουν. Ευχαριστώ. Κέλλη, ένα λεπτό. Πρόεδρε, υπερψήφισα γιατί συμφωνώ με τις προτάσεις το είπε και ο συνάδελφος σχετικά με τα ορεικτά. κάψουμε τις εκπομπές μπαίνουμε ε, προς τη σωστή κατεύθυνση και προάγουμε νέε γενναίε καυσίμων. Πολύ σημαντικό. Σημαντικό διότι εξασφαλίζει ασφαλεία δικαίου του επενδυτέ, Κρίσιμη αξία αν θέλουμε να προωθήσουμε και τα δύο καύσιμα. όλα αυτά συνάδουν με του στόχους που ανέφερε ο Επίτροπος για την Ενεργειακή Ένωση στην Ευρώπη. Τα βιοκαύσιμα βεβαίως θα διδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Είναι ενθαρρυντική λοιπόν η εξέλιξη στον τομέα της νομικής ασφάλειας, όπως είπα, της ασφάλειας δικαίου. Και γι' αυτό υπερψήφισα, όπως ε, προείπα, και εύχομαι κάθε επιτυχία στον τομέα. Για την Επιτροπή Άουκεν, μείωση χρήσης πλαστικών σακουλών. Κύριε Πρόεδρε, δίστασα για το πώς θα ψηφίσω. Δεν ξέρω κατά πόσο λύνεται έτσι το πρόβλημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν πρέπει να το αφήσουμε στα χέρια των κρατών μελών βάσει της αρχής τη επικουρικότητα. Δεν αγνώ παρόλα αυτά το γεγονός ότι είναι θεμητό ο στόχος και τελικώ υποστήριξα αυτήν την λύση. Μια λύση που θα επιτρέψει τα κρατημέλη ακριβώ να θεσπίσουν τα δικά του μέτρα προκρίνοντας τις ε, κατάλληλες κρατόπους λύσεις. Η πρόταση εν τέλει ήταν καλύτερη από την αρχική, η οποία επέβαλε στα κρατημέλη συγκεκριμένε υποχρεώσει, μεταξύ άλλων την χρέωση των σακουλών. Θεωρώ ότι η υποχρέωση αυτή δεν ήταν δυνατόν να επιβληθεί και καλύτερα κάναμε που πρόκριναμε γενικού στόχου και από εκεί πέρα τα κρατημέλη φυσικά θα την εφαρμόσουν στην πράξη. Ευχαριστώ. Μπογκοβίτσα, ένα λεπτό. Θέλω να σας πω ότι υποστηρίζω αυτή την έκθεση διότι οι πλαστικές σακούλες εμφανίζονται κατά εκατομμύρια στην Ευρώπη και ρηπαίνουν το περιβάλλον. Εμένα λοιπόν αυτό που μου αρέσει είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα με βάση την αρχή της επικουρικότητας να αποφασίσουν μόνα τους πώς θα πετύχουν το στόχο τους. Υπάρχει βέβαια μια οριακή τιμή, ένα στόχος για το έτος 2019 και το 2020. Αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι, τότε το Κοινοβούλιο θα αναγκαστεί να ζητήσει αυστηρότερα μέτρα. Μέχρι τότε όμως τα κράτη-μέλη μόνα τους θα αποφασίζουν πόσες πλαστικές σακούλες θα χρησιμοποιούν και πώς θα περιορίσουν τη χρήση τους. Επόμενος ο κύριος Νέκοβ για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ στήριξα αυτή την έκθεση γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να προστατεύουμε το περιβάλλον. Και θέλω να σας πω ότι όλοι μας ανησυχούμε γιατί καταναλώνονται πάρα πολλές πλαστικές σακούλες. Πιστεύω λοιπόν ότι παρόλα αυτά δεν είναι καλή ιδέα να επιβάλλουμε περαιτέρω κυρώσεις ε, γιατί ζούμε σε μια εποχή κρίσης ίσως αυτά να ακούγονται πολύ ωραία να χαϊδεύουν τα αυτιά αλλά έχουν και οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που δεν πρέπει να γνωρούνται. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να επιβάλλουμε ποινές ε, στους καταναλωτές που θα είναι υπερβολικά και μη ρεαλιστικά υψηλές. Εξάλλου, μην ξεχνάτε, αν ε, πάψουμε να παράγουμε πλαστικές σακούλες, θα πρέπει να απολυθούν εργαζόμενοι. Και βεβαίως, διακόπτει ο πρόεδρος, ε, επόμενη μιλήτρια, η κυρία Χάκεν. Χαρκίν, χάρηκα που ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. 92% των πολιτών μας στο Ευρωβαρόμετρο δηλώνουν ότι ανησυχούν για τις πλαστικές σακούλες και ζήτησαν να μειωθεί η χρήση τους. Εμείς στη χώρα μου ανοίξαμε το δρόμο, μειώσαμε κατά 90% τη χρήση των σακουλών. Θεσπίζοντας χρέωση για τις σακούλες. Τα σούπερ μάρκετ και οι σακούλες δεν δικούνται πλέον να χορηγούν δωρεάν. Σακούλες χρεώνουν 22 λεπτά. Είναι αρκετό το ποσό. Και έτσι οι άνθρωποι το ξανασκέφτονται στο 90% των περιπτώσεων παραλαμβάνουν οι καταναλωτέ είτε θα επαναχρησιμοποιήσουν τι σακούλε ή θα αγοράσουν ανακυκλώσιμε σακούλες. Πιστεύω ότι το σημερινό σύστημα είναι εν τέλει ευέλικτο και τα κρατημέλη μπορούν να επιλέξουν είτε να θεσπίσουν υποχρεωτικές μειώσει, είτε να θεσπίσουν κανόνε για την ανακύκλωση και την λιπασματοποίηση των σακουλών. Πέτει ένα λεπτό. Πρόεδρε, είμαι μάρτυρες του τελευταίου βήματος, μια μακρά πορεία για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι πλαστικές σακούλες καταλήγουν στη θάλασσα, στην ξηρά, εκτός του κύκλου της ανακύκλωσης. Η τρομακτική αυτή χρήση σακουλών αποτελεί απειλή. Πρόκειται για μη βιώσιμη δραστηριότητα. Πρόκειται δραστηριότητα που προκαλεί τρομακτική ρήπανση. Η οδηγία λαμβάνει υπόψη ακριβώ τι συνήθειε των καταναλωτών, τι ανάγκε των παραγωγών, αλλά και την ανάγκη μείωση τη ρήπανση. Οι αλλαγέ λοιπόν που επιφέραμε και η μείωση του πάχους από τα 15 στα 10 μικρά επιτρέπουν την χρήση των πολύ ελαφρών των πολυλεπτών σακουλών. Θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα για την μείωση τη κατανάλωσης, αλλά το καλό είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν επιλογές. Ευχαριστούμε ο κύριο Κέλλη για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ψήφισα όπως και η ομάδα μου ολόκληρη και υπέρ και χαίρομαι γιατί και η πλειοψηφία ψήφισε έτσι υπέρ δηλαδή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σοβαρό είναι το θέμα και ότι πρέπει κάτι να γίνει γι' αυτό. Καλό είναι που υπάρχει στόχος ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος. Όταν πρέπει κανείς να πληρώσει για κάτι, διστάζει να κάνει κατάχρηση του. Στη Δανία και σε άλλες χώρες λένε ότι ο καθένας χρησιμοποιεί μόνο τέσσερις πλαστικές σακούλες το χρόνο και στη χώρα μου επιβλήθηκε ένα πρόστιμο για τις πλαστικές σακούλες 15 λεπτών τώρα έχει γίνει 20 λεπτά και μειώθηκε έτσι η χρήση σακουλών από 380 την ημέρα κατά 21% πράγμα το οποίο προστατεύει το περιβάλλον. Η κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ. Και εγώ υποστήριξα τις τροπολογίες για την οδηγία για τις πλαστικές σακούλες διότι έτσι λαμβάνονται υπόψη και οι θέσει των μικροπαραγωγών της Κροατίας. Το γεγονός είναι ότι οι ελαφρές πλακτικές σακούλες είναι και αυτές βλαπτικές για το περιβάλλον, άρα η λύση είναι η ανακύκλωσή τους. Δυστυχώς όμως μια τέτοια πρόταση δεν έγινε δεκτή και η συμβιβαστική λύση που προτείνει η οδηγία είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνη. Η πληρωμή των πλαστικών σακουλών από το 18 και μετά συμπεριλαμβάνει μόνο τις πολύ ελαφρές και λεπτές πλαστικές σακούλες και ελπίζουμε ότι έτσι θα μειωθεί η μείωση η του περιβάλλοντος και γι' αυτό δέχτηκα την πρόταση. Σρόντερ ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να εξηγήσω γιατί γιατί ψήφισα όπως ψήφισα. Οι πλαστικές σακούλες οι λεπτές πλαστικές σακούλες μέχρι 15 μικρά ε, λέγονται ελαφρές πλαστικές σακούλες αλλά η οδηγία δεν συστήνει τίποτα λέει δίνει στα κράτη-μέλη την επιλογή του τρόπου με τον οποίο θα μειώσουν την κατανάλωσή τους είτε με εσωπληρωμή είτε άλλος επίσης σημειώνω ότι πρέπει να υπάρχει σήμανση για τις σακούλες που είναι βιοαναλώσιμες. Και νομίζω ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή της σε θέματα που δεν μπορεί να λύσει το κάθε κράτος και γι' αυτό υπερψήφισα. Η έκθεση Φαρία τώρα, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές. Κυρία Χάρκεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι καλή η πρόταση αυτή και σε αυτό το θέμα είναι πρωτοπόρος η Ένωση. Στόχος είναι η ισοτιμία διεθνώς. Το 4% όλων των εκπομπών διοξιδίου προέρχεται από τις θαλάσσιες μεταφορές και προβλέπεται αύξηση του. Ο Οι δομές θαλάσσιων μεταφορών είναι ο μόνος τομέας που δεν καλύπτεται από άλλες, ε, άλλα νομοθετήματα για τις εκπομπές. Άρα έπρεπε κάτι να γίνει και χρειάζεται ένα υπερεθνικό πλαίσιο. Αλλά από κάπου έπρεπε να αρχίσουμε και αυτή είναι μια καλή αρχή. Όλα τα πλοία που θα μπαίνουν, θα ελιμενίζονται σε ευρωπαϊκούς λιμένες θα την κάνουν επαλήθευση και ελέγχου για τις εκπομπές τους και από και προς ευρωπαϊκά λιμάνια και θα πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία τους. Να συλλεχθούν στοιχεία για την ενεργειακή αποδοτικότητα επίσης. Η πρόταση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τεράστιο κόστος. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κέλλη πάλι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που η σύσταση αυτή έγινε δεκτή προηγουμένως και τώρα θα γίνει επιτέλους κάτι για τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα που προέρχονται από τις θαλάσσιες μεταφορές. Όπως είπαμε και το πρωί, μέχρι 4% των εκπομπών διοξιδίου προέρχονται από τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών και κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους, ιδιαίτερα για το μέλλον. Πρέπει να επιτηρούμε, να εποπτεύουμε τα, τη δραστηριότητα των πλοίων που θα ελιμενίζονται και από εκεί και πέρα. Και πέρα μπορεί να γίνει κάτι και διεθνώς. Κάτι που θα βοηθούσε στην επίλυση του προβλήματος. προβλήματος. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και δείχνει ότι το Κοινοβούλιο και η Ευρώπη μπορούν να κάνουν κάτι για τους πολίτες τους. Ευχαριστούμε πολύ. ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην έκθεση Βαλένσα. Δίνω τον λόγο στην κυρία Χάρκιν για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Εγώ θεωρώ πως η έκθεση Βαλένσα για τις προτάσεις της Κομισιόν για ένα πολιετές ε, σχέδιο για τα αποθέματα Ρέγκας ε, και Μπακαλιάρου είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Αναφερθήκαμε ήδη και στο θέμα της αλληλείας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντέιβις για τον ρόλο τον οποίο έπαιξε για την βελτίωση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Ο ρόλος μας τώρα εδώ πέρα είναι να εξασφαλίσουμε την σωστή εφαρμογή των συμφωνημένων. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για το ότι έγινε δεκτή η τροπολογία 30 που αφορά τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα επίσης. Ε, βλέπουμε πως υπάρχει ένας δείκτης ε, θνησιμότητας ε, των αποθεμάτων που λέγεται δείκτης θνησιμότητας εντό του οποίου μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση και βεβαίως αφορά και τον γόνο και την επίδραση που έχουν τα θαλασσοπούλια και τα λοιπά θαλασσια ζώα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πετή για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο επίσης απαιτεί από τα κρατημένα να ευθυγραμμίσουν τις ε, πολιτικές τους για να διαχειριστούν με σωστό τρόπο το θαλάσσιο περιβάλλον. Τα εμπορικά είδη, αλλά και τα υπόλοιπα πρέπει να προστατευτούν για να προστατεύσουμε το οικοσύστημα αυτή τη στιγμή όταν ε, τα αλλιεύματα είναι πέραν του σημείου της αηφορίας χωρίς να σεβαστούμε μια βιώσιμη προσέγγιση δεν θα πετύχουμε τους στόχους των ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών μέχρι το 2020 ή δεν θα διατηρήσουμε βεβαίως την βιωσιμότητα αυτού του κλάδου της οικονομίας ε, που έχει σημασία για τις μελλοντικές γενιές. Περνάμε τώρα στην έκθεση Καντέκ. Ο κ. Μπόκοβιτς για ένα λεπτό σας ευχαριστώ. Εγώ στήριξα την έκθεση αυτή, την υπερψήφισα, καθώς χαλαρώνει τους κανόνες για τις υποχρεώσεις που έχουν οι αλληλείς να εκφορτώνουν σε ηχθειόσκαλες. Η πρακτική εμπειρία μας δείχνει πως υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στην εφαρμογή αυτής της οδηγίας, οπότε σύμφωνο με την ε, πρόταση πως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη σύνταξη ενός νέου εγγράφου και πρέπει να ακούσουμε και τους ψαράδες βεβαίως. Σε χώρες όπως την ε, Σλοβενία όπου εμείς εκφορτώνουμε λίγου, λίγες εκατοντάδες ε, τόνους ε, ψάρια ετησίω. Είναι μεγάλο βάρος αυτοί οι κανόνες. Και άρα εμποδίζουν και τον τουρισμό. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Την έκθεση Λιμπάτσκα. Εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνιας. Η κυρία Σόιντροβα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που δίνετε να γνωμοδοτήσω και εγώ να εκφράσω την άποψή μου για αυτή την ε, έκθεση που υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνιας. Συνετάχθη από την κυρία Λιμπάτσκα, την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω. Πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή αναλυτική έκθεση και είχαμε και καλή συνεργασία. Δυστυχώς ε, στην Ολομέλεια δεν καταφέραμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό με σωστό τρόπο και να τονίσουμε πως η έκθεση αυτή κυρίως ενισχύει τις περαιτέρω δυνατότητες ε, χρηματοδότησης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιωθεί η ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης ε, στο πλαίσιο του λεγόμενου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευση επίση. η έκθεση προετοιμάστηκε στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου του Μαΐου στο Ερεβάν και είναι ένα είδος έντολης. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεργασία. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Η μεταρρύθμιση του συστήματος της ανώτερης εκπαίδευσης ξεκίνησε με τη διαδικασία της Μπολόνια. Το θέμα είναι να δούμε ποιος είναι ο απολογισμός. Έχουμε θετικά, αρνητικά. Δεν νομίζω όμως ότι είμαστε σε θέση να πούμε. Βασικός στόχος είναι η σωστή προετοιμασία για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει γιατί η διαδικασία της Μπολόνια τελικά έχει ανατρέψει το διοικό σύστημα το οποίο επικρατούσε, το οποίο έβαζε τις ανώτατες σχολές από τη μία και τα πανεπιστήμια από την άλλη. Έχουν υπάρξει λοιπόν αντιστάσεις πάρα πολλές στη διαδικασία της Μπολόνια. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε marketing, το θέμα είναι να καταλήξουμε σε σωστές αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ. Την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια γιατί εν λόγω διαδικασία αξιοποιήθηκε προκειμένου να προωθηθεί η υπονόμευση του δημόσιου χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. έτσι άνοιξε ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση ενός καθαρά δημόσιου αγαθού όπως είναι η εκπαίδευση σε τριτοβάθμιο επίπεδο και επιβλήθηκαν τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά στα αε στην ελλάδα. η διαδικασία της μπολόνια υποτίθεται ότι θα συνέβαλε σημαντικά στην απασχόληση όμως η ανεργία των νέων βρίσκεται στα ύψη. στην ελλάδα έχει φτάσει στο 51,7 200.000 νέοι επιστήμονες δηλαδή το 2% του ελληνικού πληθυσμού μετανάστευσαν στις χώρες του σκληρού πυρήνα της ευρωπαϊκής ένωσης ταυτόχρονα η μείωση των κονδυλίων για την παιδεία που επιβλήθηκε με τα μνημόνια στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου σε συνδυασμό με τις επιταγές της μπολόνια δρομολογούν την εκπαίδευση προς μια καθαρά εμπορική προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Το βασικό μήνυμα της έκθεσης αυτής είναι ότι η διαδικασία της Μπολόνια χρήζει μεταρρύθμισης. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε το 1999 και εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες οι οποίες υιοθετούν τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης και της εμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων. Η ανταλλαγή των εμπειριών και των πρακτικών σε πανεπιστημιακό επίπεδο είναι ο καλύτερος τρόπος για τη βελτίωση της κατάστασης. Βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει κάποιες αλλαγές σε επίπεδο οργανωτικό και σε επίπεδο συγκρισιμότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων. Από την άλλη όμως υπάρχει έλλειψη επαφής και επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Σβέρκο, ένα λεπτό. Συγγνώμη, έκανα λάθο. Η κυρία Ζαμπόρσκα έχει το λόγο πρώτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συγκρισιμότητα της ποιότητας της παιδείας και η άρση των φραγμάτων δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους που μπορούν έτσι να επωφεληθούν αν ασχέτως της χώρας από την οποία προέρχονται. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω μαζί με την συγκήτρια την σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της διαδικασίας της Μπολόνια και του προγράμματος Εράσμου. Υψηλός ρυθμός ανεργίας των νέων δείχνει όμως ότι δεν πρέπει άκρητα να στηρίξουμε τις σπουδές διότι βλέπουμε ότι όσοι έχουν ανθρωπιστικές σπουδέ βρίσκουν δυσκολία να βρουν κάποια θέση εργασίας και ούτε η τεχνολογία πάντοτε σώζει. Πρέπει να βρούμε μία σύνδεση μεταξύ των αξιών. Ευχαριστούμε κύριο Σεσβέρ τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την συγκήτρια για την εξαιρετική της έκθεση ως προς την εφαρμογή της διαδικασίας της Βολονίας. Ευχαριστούμε κυρία Λιμπάτσκα. Επίσης να την ευχαριστήσω για την προσέγγιση της γενικότερα Ισκιώδης. θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο κείμενο, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο κείμενο της έκθεσης. Η διαδικασία της Βολονίας έχει πολύ συζητηθεί στην αρχή. Τα είπαμε όλα από την αρχή και πρέπει επιτέλους κάτι να γίνει. Είναι από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις η διαδικασία της Βολονίας και μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις και εκτός των συνόρων της Ένωσης. Είμαι βέβαιος ότι μπορεί έτσι να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των σπουδών και των αγώνων, αναγκών της αγοράς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα την έκθεση πρωτοβουλία την οποία παρουσίασε η συνάδελφος γιατί νομίζω ότι 15 χρόνια μετά από τη θέση σε ισχύ της διαδικασίας της Μπολόνια απαιτείται να υπάρξει ένας απολογισμός σοβαρός πλέον. Η έκθεση η οποία παρουσιάζεται σήμερα έχει πολλές ελλείψεις όχι μόνο υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τη διαδικασία της Μπολόνια λόγω των αντιμεταρρυθμιστικών πρακτικών πολλών χωρών μελών, αλλά αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στο Ιταλικό Πανεπιστημιακό Σύστημα, το οποίο κατέρευσε μετά από τις περικοπές του Τρεμόντι και μετά από τις συνεχείς πολιτικές λιτότητας. Στην ουσία αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αντικαταστήσουμε, αυτό προσπαθεί δυστυχώ η Ένωση, το πνεύμα της μάθησης και της έρευνας με το πνεύμα του ανταγωνισμού και αναιρεί το δικαίωμα στην ελεύθερη έρευνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στην επόμενη έκθεση για τον κινηματογράφο. Ευχαριστώ λέει η κυρία Σόντροβα. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη συγκεκριμένη έκθεση για τον κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή. Ο κινηματογράφος αντιπροσωπεύει μια πολιτιστική κληρονομιά αλλά και μια ισχυρή οικονομική δύναμη. Στηρίζω επίσης το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι ο κινηματογράφος είναι τόπος συνάντησης, σύγκλησης και πρέπει να στηρίξουμε και τον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε σωστά την κινηματογραφική παραγωγή και τις επιθυμίες επίσης των θεατών, των πολιτών. Η δημιουργοί δυστυχώς είναι πάρα πολύ ανήσυχοι σε σχέση με το μέλλον της δραστηριότητάς τους. Είναι μια καλή έκθεση λοιπόν η οποία υποστηρίζει και το βραβείο Λουξ. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. την έκθεση για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο γιατί οι κινηματογραφικές ταινίες είναι πολιτιστικά και οικονομικά αγαθά που συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας ενώ ταυτόχρονα θα μπορούσαν να συμβάλλουν και στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης των κρατών μελών της ένωσης παρότι η ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως εντούτοις λόγω της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας κινείται σε μια αγορά εκ των πραγμάτων κατακαιρματισμένη. γι' αυτό πρέπει να διασφαλιστεί η προώθηση η διασυνοριακή διανομή και η προσβασιμότητα που συνδυάζεται απαρέγκλιτα με την ανάπτυξη ακροατηρίου. είναι πάντως σημαντικό ότι μέσα από το πρόγραμμα media διασφαλίζεται πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης. πρέπει να διασφαλίσουμε τη λειτουργία των μικρών και ανεξάρτητων κινηματογραφικών αιθουσών ιδίως σε μικρές πόλεις και στο πλαίσιο αυτό για την ελλάδα πρέπει να προβλεφθούν πηγές χρηματοδότησης για τη λειτουργία των θερινών κινηματογράφων που αποτελούν σημαντικό πολιτιστικό κεφάλαιο για την πατρίδα μου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 neophodno je jačati europsku filmsku industriju i ovo su alarmantni podaci koji na to ukazuju te razvijati kvalitetne instrumente financiranja. imamo jedan od izvora financiranja to je program unije kreativna europa koji ima proračun od jedne i pol milijarde eura za razdoblje četrnaesta dvadeseta ali za čitavu filmsku industriju europske unije i kompletno kulturni sektor na razini europske unije. iz pod programa medija financira se razvoj novih filmova traenje partnera i promocija izvan nacionalnih granica ovaj potprogram sufinancira razvoj i distribuciju tisuu filmova godinje i drago mi je to su korisnici iz republike hrvatske uspjeli ostvariti etiri projekta. podrala sam ovo izvjee kojim se potie kreiranje pravnih okvira javnog i privatnog investiranja i promocija europske filmske industrije. hvala. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Κώστινκα για την εξαιρετική αυτή η έκθεση, εξαιρετική και για την έγκρισή της βέβαια. Εγώ υπερψήφισα. Η δασοκομεία και τα δάση είναι κάτι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα στις χώρες όπου έχουμε πολλά δάση. Η Σλοβενία είναι από τις τρεις χώρες μέλη όπου υπάρχουν τα περισσότερα δάση. Πάνω από δύο τρίτα της επικράτειάς μας είναι δάση. Και η δασοκομεία και η επεξεργασία της ξυλίας είναι πολύ σημαντικές πηγές σε βιώσιμης ανάπτυξης και για τη Σλοβενία και για την Ευρώπη γενικότερα in tudi pomen ε, Πρέπει βέβαια αυτό να συνδυαστεί με την ε, προστασία του περιβάλλοντος γιατί μπορεί και αυτές οι βιομηχανίες να χρησιμοποιηθούν με καταχρηστικό τρόπο για την... Ε, Κύριος Πόσπισιλ για ένα λεπτό σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αρχικά εγώ ήθελα να στηρίξω αυτή τη στρατηγική αλλά τελικά δεν το έκανα Τελικά απήχα. Γιατί πέρασαν κάποιες τροπολογίες της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος σύμφωνα με τη δική μου άποψη και την άποψη τσέχων ειδικών ε, υπάρχει μια προτίμηση στην περιβαλλοντική πτυχή έναντι των συμφερόντων των ιδιοκτητών των δασών που θα πρέπει να μπορούν να ζήσουν από αυτή τη δουλειά Οπότε εγώ δεν ε, στήριξα την έκθεση. Στην Τσεχία υπήρχε μια ένωση των ε, ιδιωτών ιδιοκτητών δασών και μίλησα μαζί τους. Πρέπει να βρεθεί ένα συμβιβασμός μεταξύ προστασίας του δάσους και συμφερόντων των ιδιοκτητών. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη των δασών. Ευχαριστώ. Πιτσούλα τον Ίνο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Παρά το ότι... Smatram kako bi nova strategija o šumama trebala snažno naglasiti njihovo očuvanje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 μήπως. Όλοι χωρίς μικρόφωνο. Παρά το ότι δεν είναι αρμόδια για τη δασοκομεία, ορισμένα εθνικά, δεν αρμόδια, ορισμένα εθνικά προγράμματα μπορούν να την επηρεάσουν. Πρέπει όμως να, χρησιμο, να διαχειριστεί η διαχείριση στη δασοκομεία με υπεύθυνο τρόπο και που να μην καταστρέφει το περιβάλλον αλλά να το προστατεύει. Τα παραδείγματα από την Κροατία δείχνουν ότι οι κλοπές ξυλίας προέρχονται από μία αναρμόδια λαθασμένη κατανομή δραστηριοτήτων και δικαιοδοσιών. Συχνά λέμε ότι δεν βλέπει κανείς, λέει μια δυτική παροιμία, δεν βλέπει κανείς το δάσος λόγω των δέντρων, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ισχύει είναι ότι τα κέρδη μας εμποδίζουν να δούμε το πρόβλημα. Τα δάση είναι οι πνεύμονες της Ευρώπης και πλουτοπαραγωγικές πηγές. Πρέπει να τα προστατεύσουμε. Δυστυχώς είναι ευκολότερο να δημιουργήσει κανείς ερήμους παρά δάση. Ο κύριος Μαριάς. Η δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επικεντρωθεί στη βιώσιμη διαχείριση των δασών με κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος ιδίως σε μια κρίσιμη φάση που χαρακτηρίζεται από την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο αυτό πρέπει να μειωθούν οι κίνδυνοι δασικών πυρκαγιών ιδίω μάλιστα εν ώψη τη έλευση τη θερινή περίοδου. για τον λόγο αυτό η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να στηρίξει χρηματοδοτικά την ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη τη ευρωπαϊκή ένωση για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. κύριε πρόεδρε τα δάση και η δασοκομεία διασφαλίζουν όχι μόνο καλή ποιότητα ζωή αλλά συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη στη δημιουργία θέσεων εργασία και προστιθέμενη αξία όμως η οικονομική εκμετάλλευση των δασών προκειμένου να γίνεται πραγματικά με βάση την αειφορία πρέπει να διασφαλίζεται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να έχουμε μακροχρόνιο σχεδιασμό ενίσχυση της αρχής της βιωσιμότητας και των τεχνολογιών και τήρηση των ορίων του βιώσιμου εφοδιασμού. κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την έκθεση γι' αυτό και απήχα από την ψηφοφορία. Έχει σημασία να δώσουμε βάρος στη δασική παραγωγή. Τα δάση μας βοηθούν γενικότερα και στη διατήρηση της βιοπικιλότητας, η οποία διασφαλίζει ε, πρώτες ύλες για τρόφιμα, καλλιντικά κτλ. Δεν πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε απλά τα δάση, θα πρέπει να προστατεύσουμε και το σύστημα γύρω από τα δάση. Αν βλάψουμε τα δάση τότε θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα και στο τέλος θα υπάρξει και απερίμωση των ορεινών περιοχών και δυστυχώς η τάση αυτή υπάρχει ήδη. Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τη σωστή στρατηγική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαμορφώσει και αυτή με τη σειρά της ε, μια ε, πολιτική σωστή συντήρηση των χορτολιβαδικών εκτάσεων. Μόνο με τον τρόπο αυτό ε, θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη φυτική παραγωγή στο μέλλον. Κυρία Πέτυρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ύπαρξη των δασών για ε, το ε, μέλλον και για τις ε, μελλοντικές γενναίες. Είναι απαραίτητο και για την υγεία των μελλοντικών γενεών. Τα δάση επίσης συνεισφέρουν όχι μόνο στην υγεία απευθείας αλλά ταυτόχρονα καταπολεμούν και τις συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών εν για μας ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν και η βιοπικιλότητα τους επηρεάζει άμεσα το περιβάλλον και όπως είπα την υγεία. Η Κροατία έχει μία μακρά παράδοση σωστής διαχείρισης της ε, δασικής παραγωγής και θα πρέπει ε, να χρησιμοποιήσουμε τις κοινοτικές ρυθμίσεις αλλά και τις σωστές εθνικές ρυθμίσεις. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάλετιτς, ένα λεπτό. Ο τομέας αυτός ε, της ε, δασοκομείας στην Ευρώπη απασχολεί 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Από πλευράς λοιπόν οικονομικής ε, και κοινωνικής συμμαχίας σημασίας πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα, να διαχειριζόμαστε τα δάση με τρόπο βιώσιμο και να προωθήσουμε τη βιωσιμότητά τους. η βιομάζα του ξύλου και η χρήση της ε, σημαίνει πως θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο επεύθυνοι στην διαχείριση των δασών. Εδώ πέρα λοιπόν ε, αναδεικνύεται η σημασία του τομέα αυτού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρη στα τεχνολογικά επιτεύγματα και την εμπειρογνωμοσύνη που έχουμε στην Κροατία, η Κροατία μπορεί να συνεισφέρει στην προώθηση αυτού του κλάδου και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και αυτός είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Διακόπτουμε την συνεδρίαση και αναλαμβάνουμε στις 3. Ευχαριστώ.